και θα είναι και στο μέλλον ένα σημαντικό τρόπο για να πλησιάσουν τα εθνικά κοινοβούλια στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κλείνει και αυτή η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρία σε ολομέλεια είναι αύριο στι 9 η ώρα μέχρι τι 1.30. Η μέση διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Τέλο τη συνεδρία.